παραπευθεί αυτή η αίτηση στην Νομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η δεύτερη ανακοίνωση αφορά το γεγονός ότι από την ομάδα του ΕΛΚ και των σοσιαλιστών έχουν γίνει αιτήσει για διορισμό μελών στις, σε αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Ρέσλερ για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτού και η κυρία Φραντσέσκα Μπαρούτσο για την Επιτροπή για τις Δημόσιες Ελευθερίες, την δικαστικά και εσωτερικά και επίσης στο, στην υπηρεσία για στην Επιτροπή για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις σε σχέση με αυτές τις προτάσεις, θεωρούμε ότι έχουν εγκριθεί αυτές οι προτάσεις διορισμού από την Ολομέλεια. Έχουμε λοιπόν κλείσει τα θέματα της ημερησίας διάταξης μέχρι στιγμής, οπότε μέχρι τις 12 μπορώ να διακόψω την ημερήσια διάταξη, την συνεδρίαση.